Συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Um, uh, we the two Λοιπόν, έχουμε και τις δύο επιτροπές εδώ. Καλωσορίζω λοιπόν τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ. στην αίθουσα αυτή που συζητούμε σημαντικά θέματα από το πρωί έχουμε τον Κλάδιο Μωράης, τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τον οποίον καλωσορίζω σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση. Από τις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, ο αρμόδιος είναι εδώ, ωραία, όπως και ο κύριος Κράμερ, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις θα ακούσουμε την εκτίμησή του σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θα ήθελα μάλλον αμέσως να δώσω το λόγο στον Κλάουδιο να μας ενημερώσει από τις ουσίες πού βρισκόμεθα και θα ακούσουμε τις εμπεριγνώμονες ε, μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την πρόσκληση σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και για την ε, μεγάλη συμμετοχή αυτήν την πέμπτη απόγευμα. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και επομένως να πω ότι ο πλευρός Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επανλημμένως είχαμε ζητήσει την προσχώρηση της ενώσεως ε, στη σύμβαση ε, για την καλύτερη προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των ιδιωτών. Η 2.13 απόφαση οδήγησε σε μια εξέταση ενδελεχέστερη της κατάστασης. Ο κύριος Τίμερμαν τα εξήγησε αυτά πολύ καλά ως υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη και το διάβημα στον ε, πρόεδρο Γιούνκερ ήταν σαφέστατο. Επομένως από την υλοποίηση του μνημονίου κατανόησης της 27ης Ιανουαρίου εκλήθη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις δημονετεύσεις για το σχέδιο συμβάσεως. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς λοιπόν ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για την κίνηση αυτή. Ε, περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον να ακούσω τους κυρίους Κρεάμερ και Πάσος και ευχαριστώ εκ νέου ε, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και την Πρόεδρό της για την υποστήριξή της και τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης και εγώ σας ευχαριστώ και προτού δώσω τους λόγους, ε, το λόγο με συγχωρείτε στους εμπειρογνώμονες να πω και εγώ και να επαναλάβω ότι πρέπει να μην ε, λησμονούμε ότι έχουμε και την, ε, τις επιπτώσεις που απορρέουν από την ε, γνωμοδότηση αυτή από το Συμβούλιο αλλά βεβαίω καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης μας καλεί να συνεχίσουμε την συζήτηση δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο την πτυχή αυτή. Ο κύριο Πάσο. ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας καλέσατε να σας παρουσιάσουμε, να σας υποβάλουμε μια πρώτη εκτίμηση και είναι πράγματι πρώτη και χαίρομαι που είναι και ο συνάδελφος ε, Κρέιμερ εδώ ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει προσπαθήσει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια που συζητούμε τη συμφωνία αυτή ήταν το Μάρτιο του 10 πριν από πέντε χρόνια που η Επιτροπή σας είχε διοργανώσει μια συνεδρίαση για να προετοιμαστεί ένα ψήφισμα σχετικά μια απόφαση σχετικά με την προσχώρηση αυτή. Με συνειδήσε εκείνη το Μάρτιο του 10 λοιπόν, 18 Μαρτίου, η απόφαση του Κοινοβουλίου το Μάιο του 10 ο κ. Ραμόν Αουρέγγι που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και τον οποίο ε, καλησπερίζω με εκείνο το οποίο είχε αντίκτυπο διότι και η κυρία Κουκότ του Συμβουλίου το αναφέρει συνεχώς δηλαδή είναι ένα θέμα που γνωρίζετε δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω περισσότερο το, το, το πλαίσιο και θα πάω απευθείας στην ε, τοποθέτηση δικαστηρίου του Δεκεμβρίου. Ήδη από τον Ιούνιο είχαμε κάποιες, κάποιες πρώτες ενδείξεις γιατί παρότι ο Γενικός Εισαγγελέας επρότεινε ότι το σχέδιο συμφωνίας ήταν σύμβατο προς τη συνθήκη είχε σημειώσει τυχές επί των οποίων είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις και μας έδωσε και κάποιες ενδείξεις και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο συνάδελφος ότι επ' αυτών των επιφυλάξεων της Γενικής Αγγελέως θα μπορούσαμε να επεκταθούμε περαιτέρω. να θυμίσω καταρχάς το νομικό πλαίσιο και μετά θα πάω στην ανάπτυξη της γνωμοδότησης του δικαστηρίου. Υπάρχουν 7 εμπόδια που καθορίζει το δικαστήριο. Ώστε να πει ότι η συμφωνία δεν θα ήταν συμβατή με το πρωτογενές δίκαιο. Θα τις εξηγήσω, θα εξηγήσω τα εμπόδια αυτά και ακόμα και αν μιλώ πολύ προκατακτικά το ξαναλέω, ίσως να αναφέρω και μία-δυο λύσεις που μπορεί και να είναι πιθανές. Μπορεί και να είναι Ξαναλέω ότι είναι προκαταρική τοποθέτηση. Λοιπόν, το άρθρο 6.2 καταρχάς τη συνθήκη το οποίο λέγει ότι η προσχώρηση είναι υποχρεωτική θα προσχωρήσει δηλαδή η Ένωση αλλά δεν είναι απόλυτη θα προσχωρήσει στη σύμβαση αλλά έτσι όπως αυτό θα συνδυάζεται με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται από τη συνθήκη. Το άρθρο 8 λέει ότι η προσχώρηση δεν μπορεί να επηρεάσει τις αρμοδιότητες της ενώσεω ή των θεσμικών τη οργάνων και θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει συνέχεια των κρατών μελών ως προς την προσχώρησή τους στο πρωτόκολλο και στη σύμβαση. Αυτές ήταν οι δύο διατάξεις από τον οποίο το δικαστήριο βασίστηκε στην αιτιολόγησή του. Τώρα, για, την, για το κείμενο της 18ης ε, Δεκεμβρίου του, του δικαστηρίου. Να πούμε τρία πράγματα πρωτού μπούμε στην ουσία. Παρότι ονομάζεται γνωμοδότηση, σύμφωνα με το 218 είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η σύμβαση εφόσον έχουμε αρνητική απόφαση του δικαστηρίου. Πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε ή να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Δεύτερη πτυχή. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση τα τρία θεσμικά όργανα Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν και τα 28 κράτη-μέλη όλοι αυτοί είναι υπέρ της προσχώρησης της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν. Και όλοι προασπίζονται, ενδεχομένω με κάποιες αποχρώσεις, ότι το σχέδιο της συμφωνίας, στην οποία είχαν καταλήξει οι διαπραγματευτές, είναι συμβατή με τη Τρίτον, το ίδιο το δικαστήριο ενεπλάκη τρόπον τεινά στη διαπραγματεύση, διότι ήταν το δικαστήριο με έγγραφο που υιοθετήθηκε 5 Μαΐου του 2010, έγγραφο συζήτησης, ζήτησε την προηγούμενη συμμετοχή του δικαστηρίου στη διαδικασία ώστε να γίνει αυτή αποδεκτή. Τώρα, το άλλο στοιχείο επί του οποίου το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει συμβατότητα με τη συνθήκη Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται από αυτού, αλλά είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσεως. Δεν θα υπερβώ τα 10 λεπτά, αλλά μπορεί να τα χρειαστώ και τα 10. Καταρχά, το δικαστήριο θεωρεί ότι το σχέδιο της συμφωνίας δεν εξασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ του άρθρου 53 της χάρτας και του 53 της σύμβασης. Το 52 της χάρτας το ερμηνεύει το δικαστήριο όσο ότι δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διαφοροποιήσουν το επίπεδο της προστασίας που προβλέπει στην απόφαση Μπελώνη του δικαστηρίου, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να σεβαστούν το επίπεδο της προστασίας που προβλέπει η χάρτα και δεν μπορούν να πάνε πέραν αυτού προκειμένου να αποδεχθούν την επικυριαρχία του δροϊκού δικαίου. Ενώ το 53 της συμβάσεως εξοδοτεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει, αν θέλετε, ένταση, απόκληση μεταξύ των δύο διατάξεων. Η σήμαση μιλάει για ελάχιστα επίπεδα προστασίας και η χάρτα όχι. Ποιε είναι οι επιπτώσεις, τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν να σκεφτεί κανείς μία δέσμευση, μία δεσμευτική ανακοίνωση των κρατών μελών δεν θα πάνε πέραν του επίπεδου της προστασίας αυτής εφόσον αυτό υποσκάπτει την αρχή της επικυριαρχίας του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεύτερον τώρα, δεν υπάρχει διάταξη να αποτρέψει τα κράτη-μέλη να ελέγξουν κατά πόσον άλλος συμβαλόμενος έχει πράξει το ίδιο. Και αυτό θεωρεί το δικαστήριο ότι επηρεάζει, διαταράσει την ισορροπία και επομένως και την αυτονομία του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι θεωρητικό αυτό το ζήτημα, μάλλον. Και εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μια ανακοίνωση των κρατών μελών που θα δεσμεύονται ότι θα εφαρμόσουν τη σύμβαση σύμφωνη με τους ιστορικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο εμπόδιο είναι το πρωτόκολλο 16 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ήταν έκπληξη για κάποιους από εμά που το ακούσαμε από το δικαστήριο γιατί δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Το πρωτόκολλο αυτό όμως προβλέπει ότι τα ανώτατα δικαστήρια των συμμαλωμένων μερών θα μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γνωμοδότηση επί του σεβασμού, τη συμμόρφωση δηλαδή προ τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή κάτι σαν προκατακτική διαδικασία απόφαση υπό το ε, 267 της συνθήκη. και το κατά πόσο το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να παρακάμπτει εν πάση περιπτώσει την αυτόνομη λειτουργία τη συνθήκη που είναι ένα από τους ακρογωνίους λήθους του, του οικοδομήματος Ευρωπαϊκής Σύνωσης. Τώρα εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν το 267 με αυτές τις διατάξεις προκατακτικής τοποθέτησης εφαρμόζεται πλήρως δηλαδή η ανώτατη δικαιοδοσία από την οποία θα πρέπει να ζητούμε προκατατική γνωμοδότηση όταν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα των διατάσεων δικαίου και όταν λέμε δίκαιο μιλούμε και πλέον για τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από αυτό θα απέρε ότι δεν θα χρειαζόταν η εφαρμογή πλέον του πρωτοκόλλου 16. Άρα θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει και να μπει ότι αυτό θα ήταν επαρκές. Δηλαδή ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να επιτηρεί ίσως στενότερα την εφαρμογή του 267 παράγραφος 3 της ειδίκης αλλά θα μπορούσε επίσης κανείς να φανταστεί μια δήλωση ότι στο 14 παράγραφος 16 αν ακούσαμε καλά υπό το 76 της συνθήκης θα ίσχυε. Μετά έχουμε το άρθρο 344, τέταρτο εμπόδιο της συνθήκης. Σχετικά με πιθανή διαφορά υπό την συνθήκη, για επίλυση δηλαδή τη διαφοράς εκτός από αυτή που προβλέπει η συνθήκη και λέγεται ρητά ότι η συμφωνία προσχώρησης δεν μπορεί να επηρεάσει τις διατάξεις του άρθρου 244, 344. Αλλά ότι τα κράτη-μέλη υπό το 43 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δίνανται να υποβάλουν αίτηση προς το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από μόνο του θα υποσκέπτει, υποσκάπτει τις στοχεύσεις της διατάξεως του 344. Και το δικαστήριο θα λέει ότι θα πρέπει να έχουμε ρητή εξαίρεση του 33 τελικά και όχι 43 διόρθωση διερμηνέα τη Σύμβαση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων σε σχέση με την εφαρμογή τη συμβάσεως εντός του πεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άλλη δυνατότητα που έχουμε εδώ, που δεν είναι δική μου πρόταση αλλά της κυρίας Κοκότ, είναι ότι μία δήλωση και εδώ θα μπορούσε να επαρκεί, εφόσον λέγαμε στη δήλωση αυτή ότι τα κράτη-μέλη λένε και δεσμεύονται προς τους άλλους συμβαλωμένους της ε, Συμβάσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μην προσφύγουν ενώπιον του Ανθρωπίνου Δικαστηρίου υπό το 43 εφόσον αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Πέμπτο εμπόδιο. Εξόχως τεχνικής φύσεως γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει κράτος μέλος που να προσφεύγει στο Δικαστήριο ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων κατά άλλου κράτους μέλους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό για το 4 το 5. Ο αντίστοιχο μηχανισμός. Το δικαστήριο εδώ καθορίζει, μιλάει για δύο προβλήματα. 3F, 3F του σχεδίου Συμφωνία που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος θα πρέπει να δικαιολογεί την συμμετοχή τους στη διαδικασία και από εκεί και πέρα το Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να αποφασίζει το επαρκές το αποδεκτό της αιτιολόγησης αυτής. Και αυτό πλέον θα είναι δεσμευτικό για την Ένωση και για τα θεσμικά της όργανα εκ των οποίων και το δικαστήριο. Σχετικά λοιπόν με την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και τον αντίστοιχο μηχανισμό, δηλαδή την κοινή ευθύνη, εφόσον έχουμε κοινού κατηγορούμενους, και τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπίζονται τις αρχές του ερωικού δικαίου, αλλά μόνο ένα εξ αυτών θα είναι υπεύθυνο για τυχόν παραβίαση. Και το δικαστήριο λέει ότι μια τέτοια απόφαση του, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα σήμαινε ε, αξιολόγηση στην ουσία εκτίμηση των βασικών διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου εφόσον αυτό θα ήταν μη συμμορφούμενο προς την αυτονομία του ευρωπαϊκού δικαίου. Και το δικαστήριο λέει ότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τέτοιου είδου διαφορών. Και ότι αυτό δεν είναι ή στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιθανή λύση για το εμπόδιο αυτό σε δύο φάσεις δόσεις. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την αναδιαπραγμάτευση της ε, συμφωνίας της συμβάσεως προσχώρησης γιατί στο 35 άρθρο του σχεδίου ίσως να ήταν καλύτερο να διαγράψουμε τον όρο plausibility και ίσως και να διαγράψουμε και τη δυνατότητα ευθύνης από πλευρά ενό εκ των Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτη-μέλη. Επομένω, εδώ ίσω να χρειαστεί διαπραγμάτευση. Αυτό αφορά και στη διάταξη 37. Έκτο εμπόδιο. Διαδικασία για την πρώτερη συμμετοχή του δικαστηρίου. Και εδώ υποτίθεται το δικαστήριο απλώς εξετάζει μόνο το κατά πόσον ισχύει το παραγωγό δίκαιο και για την ερμηνεία μόνο του πρωτογενούς δικαίου, αλλά όχι την ερμηνεία του παραγωγού δικαίου. Το δικαστήριο λέει ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο. Θα μπορούσε δηλαδή το δικαστήριο θεμελιωδών δικαιωμάτων να οδηγήσει σε ερμηνεία του παραγωγού δικαίου, το οποίο θα σήμαινε ότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί τη ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου τελικά. Εδώ πρόταση πιθανής λύσεως. Αναδιαπραγμάτευση της επεξηγηματική εκθέσεως στην παράγραφο 66 και συμπερίληψη της λέξεως interpretation σε αυτή την ανάλυση. Και πάω στο πιο δύσκολο, το έβδομο, το τελευταίο. Την δικαστική επανεξέταση σε θέματα CFSP. Και εδώ πρέπει να πω ότι με εκπλήσει η τοποθέτηση του δικαστηρίου. Το Κοινοβούλιο είχε πει στο ψήφισμά του ότι αυτό ήταν η πιο απτή προστεθέμενη εξία. Γιατί το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει την ομότητα κενών που έχουν υιοθετηθεί υπό την CFSP. Αντίθετα, το δικαστήριο λέγει ότι η αρμοδιότητα προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε επανεξέταση πράξεων και υπό το φως των θεμελιωδών δικαιωμάτων και παραθέτω δεν μπορεί να παραχωρείται αποκλειστικά σε διεθνές δικαστηρίο το οποίο δεν εμπίπτει στο δικαιοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγει το δικαστήριο ε, ότι επομένως το σχέδιο συμφωνίας δεν, μπορεί, δεν σέβεται τα ειδικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με πράξεις ή παραλήψεις σε, σε θέματα CFSP. Αυτό το ανέφερε ένας μελετητής ως καταστροφικό πρόβλημα και ίσω να είναι και καταστροφικό και ω προ τη λύση που πρέπει να βρούμε. Υπάρχει τόσο ανυπέρβλητο. Εδώ η τοποθέτηση της κυρία Κοκότ ήταν απολύτως διαφορετική. Μα είπε ότι το δικαστήριο δεν είχε κανένα είδου ε, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα για θέματα CFSB. Και είπα αλλά ότι εν πάση περιπτώσει η αποτελεσματικότητα της προστασίας των πολιτών θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμωνόταν έχοντας την εξωτερική, τον εξωτερικό έλεγχο αν θέλετε του δικαστηρίου θεμελιωδών δικαιωμάτων υποθέματα ΚΕΠΑ. Εδώ δυσκολεύομαι να σας προτείνω λύσεις. Δεν ξέρω αν ο συνέδριος της Κομισιόν θα μπορέσει. Γιατί αυτό είναι πραγματικά το πιο αμφίσιμο, το πιο δύσκολο σημείο από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εδώ κλείνω. Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση είναι δύσκολος και σίγουρα θα ήταν σοφό και φρόνιμο να έχουμε μία περίοδο εξέταση σκέψης Το Κοινοβούλιο σίγουρα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και πάντα είχε σε αυτό το φάκελο, αλλά προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζουμε πλήρως ποια είναι η θέση της Κομισιόν, πώς αντιδράει η Κομισιόν προς την τοποθέτηση του δικαστηρίου. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν φρόνιμο το δικαστήριο αυτή τη στιγμή να υιοθετήσει θέση μέχρι ότου τα πράγματα γίνουν λίγο σαφέστερα εντό τη Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κρέμερ φαντάζομαι έχει κάτι να πει. Και βεβαίω. Ε, εντάξει, το κοινοβούλιο μπορεί να μην ξέρει, αλλά η Κομισιόν ε, φαντάζομαι ξέρει τι να κάνει για την ε, δήλωσή σας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε στην κοινή σας αυτή συνεδρίαση όσον αφορά το περιεχόμενο και την ανάλυση της ε, γνωμοδότησης ε, συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπε ο αγαπητός φίλος ε, Ρικάρντο Πάσος η γνωμοδότηση αυτή είναι μακροσκελής και περίπλοκη μια απόφαση την οποία ακόμα αξιολογούμε σε τεχνικό επίπεδο. όλα αυτά, ήδη από τώρα μπορούμε να πούμε πως η γνωμοδότηση απαιτεί να επαναδιαπραγματευτούμε το σχέδιο ένταξης σε κάποια σημεία. Δεν επιθυμώ γιατί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε μια λεπτομερή συζήτηση για το ποια είναι αυτά τα σημεία, αλλά να πω απλά μια τάση που υπάρχει. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος όσο ο συνάδελφος Ρικάρδο Πάσος πως ε, σε όλα τα σημεία στα οποία θεωρεί ότι αρκεί μία δήλωση ε, όντως αυτό συμβαίνει για να ξεπεράσουμε τις αντιρρήσεις ε, του δικαστηρίου. Γεγονός είναι πως ε, πιθανόν δεν είναι ε, ο, και τα 7 σημεία, πολλά από τα οποία έχουν υποσημεία, που χρειάζονται επαναδιαπραγμάτευση, αλλά ένας μεγάλος αριθμός τους όντως απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση. Είτε του διατακτικού κειμένου του σχεδίου συμφωνίας είτε του προημίου ε, προφανώς η Κομισιόν σέβεται πλήρως ε, την ε, γνωμοδότηση του δικαστηρίου και σας διαβεβαιώ πως η Κομισιόν παραμένει βεβαίως δεσμευμένη για την ένταξη της Ένωσης στην Σύμβαση. Είναι πρώτη μας προτεραιότητα και ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο πρώτος αντιπρόεδρος Τίμερμανς προσωπικά είναι δεσμευμένοι για αυτό η ένταξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση των θεμελιωδών αξιών, θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και παραμένει και δεν έχουμε αλλάξει άποψη κορυφαίας συστημικής σημασίας ε, και επιπλέον στο άρθρο 6.2 του ε, της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια νομική υποχρέωση να αναζητήσουμε μια κατάληξη σύμφωνη με αυτά τα οποία αναφέρονται στη συνθήκη και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο 8 της συνθήκης της Λισαβόνας αυτή τη στιγμή και δεδομένου του αριθμού και βεβαίως της βαρύτητας ε, των αντιδράσεων του ΔΕΚ πρέπει να υπάρξει μία περίοδος περίσκεψης για να εξετάσουμε τι θα κάνουμε από και μπρος. Και είναι σαφές πως αυτά τα οποία αναφέρει το δικαστήριο έχουν διαφορετική θα έλεγα βαρύτητα. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν κάποια νομοτεχνικά ζητήματα που αφορούν το μηχανισμό, την πρώτερη εμπλοκή του δικαστηρίου, όπως το 344 η προστασία γενικώ ε, των κανονισμών της Ένωσης από παρεμβολές του συστήματος του Στρασβούργου αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ε, είναι πολύ πιο πολύπλοκα νομικά και πολύ πιο ευαίσθητα πολιτικά. Όπως η ΚΕΠΑ, συμφωνώ εδώ πέρα, συμφωνώ με τον Ρικάρντο Πάσος, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και το πώς συνδέεται αυτό με το ότι η διαδικασία στο δικαστήριο του Στρασβούργου πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά για να βρούμε λύσεις οι οποίες θα στέκουν νομικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτι της δουλειάς μας ως Κομισιόν Κάτάχουμε ναι, κατά νου. Επίσης θα ήθελα να πω από θεσμική σκοπιά πως ε, η Κομισιόν έχει την εξουσιοδότηση από την απόφαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2010 να συνεχίσει τις ε, διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος ε, και με τα 47 και τα 47 μέλη δηλαδή τα κράτη-μέλη και οι υπόλοιποι παρακολουθούν την διαπραγμάτευση και θα συνυπογράψουν για τη συμφωνία και επίσης είναι σαφές πως στις διαπραγματεύσεις αυτές οποιασδήποτε αλλαγές ζητήσει η Ένωση θα πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα για να ικανοποιήσουμε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας ένταξης που προκύπτουν από τα πρωτοκόλλα Α έως 13. Όσον αφορά την διαδικασία, ε, οι διαπραγματεύσει θα γίνουν ε, σε συνεννόηση με την Ειδική Επιτροπή που όρισε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 2.18 της Συνθήκης ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως θα το κρατάμε ενήμερο διαρκώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ραμόν Χαουρέγγι. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ θερμότατα και στους δύο νομομαθείς πολύ διαφωτιστικές πληροφορίες που μας έδωσαν. Θα ομολογώ όμως ότι αισθάνομαι κάποια απαγοήτευση και κάποια ματέωση από το όλο θέμα. Γιατί θυμάμαι ότι το 2009 η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έδωσε αυτό το ζήτημα γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδινε τη σχετική εντολή. Ξεκινήσαμε τις εργασίες όπως είπε ο κύριος Πάσος και καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα. Βέβαια ήταν πολύ χρονοβόρα η διαπραγματευτική διαδικασία και το καταλαβαίνω, τέσσερα χρόνια για να επισημοποιηθεί η προσχώρηση. Και τώρα βλέπουμε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου που μας δημιούργησε την αίσθηση ότι ουδέποτε δεν θα υλοποιηθεί τελικά αυτή η προσχώρηση. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Άκουσα τον εκπρόσωπο της ε, νομικής υπηρεσίας που είπε σχεδόν όλα τα σημεία, όλα τα προβλήματα, όλα τα 6-7 εμπόδια που επισήμανε ε, δεν είναι ανυπέρβλητα. Ε, με δήλωση του Συμβουλίου ή με δήλωση των κρατών μελών. Εγώ θεώρησα ότι τα πρώτα έξι ε, εύκολα θα τα επιλύαμε. Το έβδομο όμως με προβλημάτισε και με θορύβησε ακόμη περισσότερο η ανησυχία του κυρίου Κράμερ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λέει δεν θα είναι εύκολο με δηλώσει να τα λύσουμε όλα. Ε, έχει την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε από την παρέμβαση του κυρίου Κράμερ, ότι έχει την αίσθηση ότι θα είναι ανέφικτη η υπέρβαση αυτών των εμποδίων. Και η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικής οντότητας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δύο νομικές συνέπειες. Καταρχήν δίνει νομική προσωπικότητα και πολιτική στην Ένωση ως ξεχωριστή οντότητας γιατί το σύνολο των 28 χωρών μελών δεν προσχωρούν από μόνα τους αλλά ως Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ως ε, νομική οντότητα προσχωρεί, αυτό έχει μια συγκεκριμένη συμβολική αξία και ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι πολίτες αποκτούν περισσότερα και καλύτερα δικαιώματα γιατί πλέον κάθε πολίτης για δράση όχι της ε, πατρίδας του αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να πλήττει τα δικαιώματά του θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δύο συνέπειες μιας πιθανής προσχώρησης. Εγώ προτιμώ μια κακή συμφωνία από την έλλειψη οποιασδήποτε συμφωνία και σας το λέω ειλικρινά. Και μια και η απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι δυνατόν να, να εφαρμοστεί, προτιμώ να αναδιαπραγματευτούμε την συμφωνία με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τη σχετική απόφαση, αλλά κάποια στιγμή να προσχωρήσουμε, όσο και να αλλάξουμε τη συμφωνία. Πρέπει να είμαστε συνετοί και να προχωρήσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπογραφεί τελικά συμφωνία για να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, βλέπω να ζητάει άλλος κανείς το λόγο. Έχω μία ερώτηση. Υπήρξε κάποια στιγμή που επίσημα το Συμβούλιο ήταν θετικό για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, και στήριξε την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση. Γιατί είναι η πρώτη απόφαση, πρώτη γνωμοδότηση τόσο αρνητική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπω είχαμε και στο παρελθόν κάποιες ε, αρνητικές ενδείξεις. Γιατί δεν ξέρω ποια ήταν η διαδικασία, πότε είναι πλάκη ε, το δικαστήριο. Στην ε, προκαταρκτική φάση των διαπραγματεύσεων είχε γνωμοδοτήσει το ΔΕΚ ή όχι. Ναι, να σας απαντήσω και θα με συμπληρώσει ο κύριος Κράμερ το ΔΕΚ ως θεσμικό όργανο ουδέποτε δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών. Γι' αυτό και είπα ότι είναι ε, περίεργο και πραγματικά εξαίρεση που το δικαστήριο υιοθέτησε ένα έγγραφο συζήτησης στις 5 Μαΐου του 2010 στο οποίο αποσαφήνισε την ανάγκη ε, ύπαρξη ενός μηχανισμού πρώτερης συμμετοχής του δικαστήριου. Χωρίς να δίνει διεξοδικές λεπτομέρειες, είπε ότι το δικαστήριο θεωρεί ως εκτορών ουκάνευ προϋπόθεση την πρώτερη συμμετοχή του στη διαδικασία. Δεν νομίζω όμως ότι το δικαστήριο συμμετείχε, ενημερώθηκε, είχε οποιαδήποτε επαφή με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και μας εκπλήσει ότι για κάποιες πτυχές της, ε, του σχεδίου συμφωνίας το δικαστήριο εντόπισε 7 παραγράφους που θεωρούσε αντιφατικές με το πρωτογενές δίκαιο. Και είναι ευνόητη αλήθεια του δικαστηρίου με το, πρωτόκολλο, με το πρωτόκολλο 16 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έκρινε ότι αυτό το πρωτόκολλο επηρεάζει το μηχανισμό των προδικαστικών ζητημάτων και των προδικαστικών αποφάσεων. Ε, εγώ το είχα φανταστεί, το είχα προβλέψει ότι θα υπάρχει πρόβλημα με το πρωτόκολλο 16 και επιβεβαιώθηκε. Τώρα για την ΚΕΠΑ έγιναν πολλές συζητήσεις για το τι θα έπρεπε να κάνει το δικαστήριο και νομίζω ότι η επιχειρηματολογία της Γενικής Αγγελέως ήταν ότι μερικές φορές ε, προβλημάτιζε ε, ενώ προβλημάτιζε η ιδέα, τελικά είναι πιο θετική για το, για το κρίσιμο αυτό ζήτημα της ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. στο μέλλον. Τι σχέδια υπάρχουν για προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη σύμβαση ή παρόμοια εμπόδια θα αντιμετωπίσουμε και στην ενδεχόμενη ε, προσχώρηση και σε άλλες συμβάσεις. Γιατί είχαμε αυτό το αυτή τη συζήτηση και την ευκαιρία τη συντακτική συνέλευση, ότι με το Σύνταγμα δηλαδή θα δώσουμε νομική προσωπικότητα στην Ένωση και ότι θα μπορέσει ε, αυθυπόστατα να προσχωρήσει στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μας ε, απογοητεύει ε, τρομερά βέβαια αυτή η αδυναμία προσχώρησης, γιατί όπως είπε και ο Κλώτο Μωράες, ε, ε, θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να προχωρήσετε. Βέβαια ψήφισμα δεν πρόκειται να συντάξουμε. Περιμένουμε την έκβαση ε, αυτής της περίοδου περίσκεψη και στοχασμού για να δούμε πώ θα ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Αλλά αν ε, βαγίσει όλη η διαδικασία, τότε η ματέωσή μας ε, θα φτάσει στο να δίρκει η απογοήτευσή μας. Φαντάζομαι ότι καλύπτω και την νομική υπηρεσία με αυτή την ε, διαβεβαίωση ότι μπορεί να περιμένει την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να σχολιάσετε, απλώς σας διαβεβαιώ ότι θα σας υποστηρίξουμε πλήρως. Και ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε, γιατί πολλές φήμες ακούγονται αριστερά και δεξιά για το τι συνέβη και πώς αν μου επιτρέπετε μια λέξη. Πρώτα απ' όλα δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα με τις άλλες διεθνείς συμφωνίες. Γιατί εδώ πέρα δημιουργείται ένας εξωτερικός ε, έλεγχος, ε, ακούστηκε ακόμα και η λέξη υποταγή, η οποία δεν είναι σωστή βεβαίω. του ΔΕΚ στο, στο Τώρα η Κομισιόν πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Πρέπει να κάνουν μια πρόταση στο Συμβούλιο για να αναθεωρηθούν οι διαπραγματευτικές οδηγίες, θα μας δώσουν ένα αντίγραφο, βεβαίως ε, αυτοί θα διαλέξουν τη στιγμή, αλλά μέχρι τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Μια προφανής ερώτηση. Πόσο καιρό θα χρειαστεί αυτή η περίοδος σκέψης της ε, Κομισιόν. Προς ε, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν απευθύνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω αυτή τη στιγμή ακριβείς ε, ενδείξεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αλλά σας διαβεβαιώ και πάλι πως εργαζόμαστε σκληρά πάνω στο θέμα. Είναι προτεραιότητα της Κομισιόν σε πολιτικό επίπεδο και βεβαίως ε, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη της, ε, την νομική πολυπλοκότητα που αποκαλύπτει η, ε, που αποκάλυψε αυτή η γνωμοδότηση. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας ε, ε επίσης κυρία Πρόεδρε, αλλά να σας θυμίσω πως την πρώτη του γνωμοδότηση το δικαστήριο την 2.94 όταν έπρεπε να εξετάσει το ζήτημα του εάν υπήρχε νομική βάση στην προηγούμενη συνθήκη που δεν υπήρχε είπε πως η ένταξη στη συνθήκη ε, έχει συνταγματική σημασία για τις ευρωπαϊκές κοινότητες όπως ήταν τότε. Τέτοιο βήμα λοιπόν συνταγματική σημασίας ε, ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο και τώρα ακριβώ είμαστε σε μια φάση όπου λόγω αυτή τη γνωμοδότησης ε, πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά για να γίνει το βήμα αυτό σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, δεν θυμάμαι πότε ήταν, μέσα της δεκαετίας του 90 το δικαστήριο είχε πει πως η κοινότητα δεν, δεν μπορεί να προσχωρήσει στην συνθήκη. Αλλά είπαν στην ίδια απόφαση πως έχει συνταγματική σημασία. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ε, ακριβώς αυτό ήταν. Σας διάβασα μέσα από την απόφαση. Ε, τώρα βεβαίως ε, έχουν διαφορετική άποψη, αλλά το γεγονός ότι έχει συνταγματική σημασία παραμένει. Ωραία, σας ευχαριστώ. Θα συνεχιστεί ο αγώνας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Λίγη η συνεδρίαση.